πάνω λοιπόν στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να δώσω τον λόγο στην Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, καλημέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και χαίρομαι γιατί με αυτή την ευκαιρία θα συζητήσουμε την ε, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη. Επίσης, στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Ισότητα των Φίλων του 2015 έχουμε ε, το ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια νομική υποχρέωση που απορρέει από τι συνθήκε και είναι κάτι που ξεκίνησε από την αρχή τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι κοινωνίε μα έχουν σημειώσει τεράστια πρόεδρο την τελευταία έξι κονταετία. Η θέση των γυναικών έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έχουν περισσότερη πρόσβαση ε, τώρα οι γυναίκε σε όλο περισσότερο από πριν και αναμφίβολα κινούμεθα προς τα εμπρός αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν πάρα πολλές ανισότητες ακόμη παρ' όλα αυτά εάν ε, συνεχίσουμε έτσι πρόκειται να μας πάρει άλλα 70 χρόνια για να πετύχουμε την ισότητα των δύο φίλων. οι γυναίκες ε, κερδίζουν 10% λιγότερα από τους γυναίκες, τους και ε, επίσης ε, μία ώρα την ημέρα ε, περνάνε με τα παιδιά τους οι πατεράδες ενώ οι μανάδες τρεις ώρες οπότε θα πρέπει να μπορέσει να συνδυάσει η γυναίκα τον ιδιωτικό βίο με τον επαγγελματικό βίο οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ανεξαρτησία την κοπική της γυναίκας δεν θα πρέπει να οδηγηθεί σε κάποια φτώχεια εάν δεν υπάρχει άλλο στην οικογένεια που να εργάζεται, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις συντάξει τι θα πρέπει να γίνει με τον ε, κίνδυνο του να πέσει σε φτώχεια γυναίκα στα γεραματά τη. Γιατί έχουμε στι συντάξεις μια ανισότητα, 40% λιγότερο έχουν οι γυναίκες και δεν υπάρχει δυστυχώ σημάδι ότι γεφυρώνεται αυτό το χάσμα. Θα πρέπει να δούμε επομένω ποιε είναι θετικέ άλλαγε των περσμένων δεκαετιών, τόσο ώστε να δημιουργήσουν μια κοινωνία όπου ε, κάθε γυναίκα ή άντρα να μπορούν να προοδεύσουν. Να σταθώ τώρα σε τρει άξονε που θα μπορούσαμε να μα οδηγήσουν σε πιο πολλή ισότητα. Οι γυναίκε είναι το μισό και παραπάνω από τον πληθυσμό. Αλλά στι περισσότερε διευθυντικέ θέσει έχουμε πιο πολλού άντρε παρά γυναίκε και επίσης στα εθνικά κοινοβούλια έχουμε περισσότερους άνδρες από γυναίκες. Αυτό αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις μεγαλύτερες εταιρείες ε, που έχουν έδρα στις ε, χώρες μέλη, 30% και λιγότερο στα διοικητικά συμβούλια είναι γυναίκες. Οπότε εμείς προτείνουμε να προχωρήσουμε προς μια εξίσωση, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή αυτή την ανισότητα και έτσι τα διοικητικά συμβούλια να έχουν τουλάχιστον 40% ε, από ε, γυναίκες. Οπότε θα πρέπει αυτό να επιβληθεί, θα πρέπει να, να, το εφαρμόσουν για τα κράτη-μέλη που ακόμα είναι διστακτικά. Θα πρέπει επομένω οι Ευρωπαίοι να συνδυάσουν τις επαγγελματικέ επαγγελματικές υποχρεώσεις με τις οικογενειακές. Κάποια στιγμή φέτος πρόκειται να παρουσιάσουμε μια δέσμη νομοθετικών και μη μέτρων, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη ισότητα για τους εργαζομένους. Θα πρέπει να εξετάσουμε στα πλαίσια εκείνα το πώ θα έχουμε περισσότερη ποιότητα στη φροντίδα των παιδιών, τι θα, θα μπορέσουν αυτοί που φροντίζουν τα παιδιά, είτε είναι πατέρες είτε μητέρες, να έχουν περισσότερη ευελιξία. Και επίσης έτσι θα βοηθήσουμε στο να ενταχθούν καλύτερα οι γυναίκε στην χώρα ε, εργασίας. Αυτό και δημογραφικά και οικονομικά είναι σημαντικό. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε και μια στην οικονομική ανάπτυξη τη Ευρώπη. Τελικά ε, έχουμε βία μεταξύ των ε, δύο φίλων. Δηλαδή, μία στις τρεις γυναίκες θεωρείται ότι έχει υποστεί ε, επίθεση η σεξουαλική, η απλή επίθεση και τις δύο. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προσχώρηση στην ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι μια συμφωνία δεσμευτική, η πρώτη, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί αυτή η διέγρα των γυναικών. Αυτή η προσχώρηση στη συμφωνία της ε, Κωνσταντινούπολης είναι το κλειδί για να προχωρήσει η στατική μας δέσμευση. Οπότε έχουμε θέλουμε μια τέτοια συνολική προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο. Αυτή είναι η ενωσιακή προσέγγιση. Οπότε ε, θεωρούμε ότι με αυτή τη συνθήκη θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και θα μπορέσουμε να δράσουμε κατασταλτικά αλλά και προληπτικά για τη βία κατά των γυναικών. Επίσης θα πιάσουν περισσότερο τόπο οι κοινοτικοί πόροι. Αυτό πρόκειται να αναβαθμίσει την αξιοπιστία μας ε, αλλά επίσης και την ε, υποχρέωση λογοδοσίας. Επίσης πρόκειται να προωθηθούν οι ευρύτεροι στόχοι κατά των δυσμενών διακρίσεων, οικονομικής ανάπτυξης και συνεργάζομαι με την Επίτροπο κυρία Τάισεν, ε, με την ε, υπηρεσία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχουμε έρευνες από την Eurostat και επομένως πρόκειται να εντάξουμε αυτές τις στατιστικές έρευνες στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα ε, που θα καλύψει τα έτη 2016-2019 εντοπίζει το ότι αυτά τα ζητήματα που αναφέραμε είναι ζητήματα προτεραιότητος και θέλουμε ισότητα των φύλων αλλά και ισότητα στην οικονομική ανεξαρτησία. Αυτού του είδους επομένως αυτή η στράτευσή μας ε, θέλουμε να καλύψει το ότι η ισότητα πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε μας πολιτική στην ε, χάραξη της πολιτικής, στην εφαρμογή, στην εποπτεία, αλλά και στην αξιολόγηση αυτών των πολιτικών και στα νομοθετικά μέτρα, αλλά και στα προγράμματα που χρησιμοποιούν κοινωτικούς πόρους. Εν κατακλείδευτα θα θέλω να σας τονίζω ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γυναικών, αλλά και το φρένο που πρέπει να μπει στην βία των γυναικών είναι κορυφαίες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Λεγκρίπ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, για τα λόγια σας που δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η προσήλωσή σας και η στράτευση και πολιτική και προσωπική προσωπικά εσείς αλλά και ως Επίτροπος αρμόδια για θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Κάνατε κάποιες διευκρινήσεις, μας δώσατε κάποια στοιχεία και διατρανώσατε και πάλι τις μεγάλες ε, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μιλώ εξ ονόματο τη ομάδα μου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, στη Παγκόσμια ημέρα τη Γυναίκα. Δύο είναι μεγάλε προκλήσει. Βελτίωση τη κοινωνικο οικονομική κατάσταση των γυναικών. Αυτό είναι ένα θέμα και ισότητα και ανταγωνιστικότητα, αλλά και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη επαναλαμβάνω, μεταξύ ανδρών και γυναικών βελτίωση της οικονομικής κατάστασης ε, της Υπήρου γι' αυτό λέω ανταγωνιστικότητα, για να καταπολεμήσουμε αυτή τη τεράστια απώλεια, γιατί πάει χαμένο το ε, ανθρώπινο δυναμικό, το γυναικείο δυναμικό, γιατί δεν έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί. Οι γυναίκες είναι εξίσου μορφωμένε, εξίσου καταρτισμένε με τους άνδρες και είναι κρίμα να χάνουμε και ανθρώπινο δυναμικό και δυναμικό γενικότερα. Γιατί δεν δίνουμε στις γυναίκες την πλήρη θέση που του αξίζει και ε, όλες τις ευθύνε ε, στην αγορά εργασία. Εμεί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανησυχούμε βαθύτατα και θα εργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες επ' αυτών των θεμάτων με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, τι μπορούμε να προτείνουμε και τι μπορεί να εφαρμοστεί. Βέβαια, μετά από πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, αλλά καλούνται και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του για να μειώσουν τι μισθολογικέ ανισότητε και τι συνταξιοδοτικέ. Ε, ε, gender pay gap και pension pay gap λέγεται αυτό στα αγγλικά ε, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι δύο μεγάλα θέματα και θα πρέπει σύντομα να επιτευχθεί πρόοδο στου επόμενου μήνε. Σα ευχαριστώ. Κυρία Λεγκρίπ, έχετε μπλε κάρτα. Ο κύριος Λαβριού θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε, βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα κάνω την εξής ερώτηση στη συνάδελφο Κωνσταντ Λεγκρυπ. Φρονείτε ότι θα ήταν ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 28 κρατών μελών να ε, υιοθετηθεί ο νόμος Κοπέ Τσίμερμαν, ε, ο γαλλικός νόμος για το 2017 θα μπορούσαμε ε, να καθιερώσουμε την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, ισομερή εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών για να προωθηθεί η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και στην ηγεσία του οικονομικού γίγνεσθεν. Μάλιστα, βεβαίω. προφανώς. Πρόσφατες μελέτε έχουν καταδείξει ότι όταν υπάρχουν τέτοια νομοθετικά κίνητρα και ισχυρά, ε, όχι μόνο για ισομερή εκπροσώπηση, αλλά για γενικότερα ισχυρότερη παρουσία ε, των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών, αυτό είναι θετικό και ευνοϊκό. Όχι μόνο για τα ίδια τα διοικητικά συμβούλια, αλλά συμπαροσύρονται και τα υπόλοιπα όργανα λήψη αποφάσεων και θα ήθελα να ε, εξάρω την προσπάθεια της κυρίας Γιώροβα για, το σχέδιο οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία πριν από μία διετία περίπου. Και η δική μας ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αγωνίζεται πάρα πολύ στεναρά προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως και χρειάζονται ευρωπαϊκά νομοθετικά ε, μέσα για να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρείων. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε, παρακαλώ. Ε, Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν από το βάθος της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω γιατί μας παρουσίασατε σήμερα το ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες από τις οποίες ζουν οι γυναίκες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι Υπάρχει ένας ε, μεγάλος ε, συμβολισμός ε, και ένα μήνυμα που παίρναμε σήμερα γιατί 8 Μαρτίου συζητάμε την κατάσταση των γυναικών και την ισότητα των γυναικών στην Ολομέλεια. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλή επιτυχία και να ζητήσω εμείς να εγκρίνουμε την νομοθεσία που ε, ευνοεί τις γυναίκες όχι μόνο κάθε 8η Μαρτίου αλλά πιο συχνά για να βελτιώσουμε την κοινωνική και την οικονομική κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι γυναίκες μπορούν να συμφιλιώσουν τον εργασιακό και τον οικογενειακό βίο. Γιατί μην ξεχνάμε πως ακόμα και στον 22ο και στον 23ο αιώνα το βάρος αυτό ε, το υπομίζονται οι γυναίκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε οι γυναίκες να χάνουν τη θέση στις εργασίες τους επειδή χρειάστηκε να φροντίσουν μέλη της οικογένειάς τους και στο κάτω-κάτω θα έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για να φροντίσουν τη δική τους υγεία οι γυναίκες. Τι γίνεται με την νομοθεσία περιγονικής άδειας ε, μητρικής, πατρικής ε, κτλ. Τι συμβαίνει με την άδεια για την φροντίδα των ηλικιωμένων συγγενών. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή θα προσφέρεται χωρίς να χάνει κανείς την ε, ε, θέση του. Πότε θα πετύχουμε τους στόχους της Βαρκελόνης έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετές θέσεις για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους και νομίζω ότι ε, χρειαζόμαστε και κάποια ψηφίσματα που θα επιτρέψουν ε, στους ανθρώπους να συνδυάσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική του ζωή. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία το σχετικό νομοθετικό πακέτο από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Φωνστόρχ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί συζητούμε την κοινωνικο-οικονομική παρακαλώ κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι κατέστησε σαφές ότι δεν είναι στο πλευρό των γυναικών που είναι μητέρες και στην οικογένειά τους. Αρνείται και εξακολουθεί να αρνείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ε, τη συνεισφορά των μητέρων στην εθνική οικονομία. Ο Κέρμπεκερ κέρδισε βραβείο Νόμπελ με τέτοια μοντέλα για το πώς δημιουργείται αξία στην οικογένεια και οι γυναίκες να αναδειχθούν. Και ο ΩΣΑ το έχει ήδη ε, αναδείξει και αναγνωρίσει όπως και τα Ηνωμένα Έθνη. Οι οικογένειες παράγουν υπεραξία και οι γυναίκες και οι μητέρες αποδίδουν, εργάζονται στο σπίτι και αυτό είναι σκληρή πραγματικότητα και δεδομένο οικονομικό. Κυρίες και κύριοι, η παραγωγή αξίας αρχίζει όταν αρχίζουμε να εκτιμούμε τις αξίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να εκτιμήσει τις γυναίκες και τις μητέρες στην οικογένεια γιατί δεν αναγνωρίζει την ε, παρουσία τους και την προσφορά τους. Μήπως να αρχίσουν σιγά σιγά. Ευχαριστώ κυρία Μπεθέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Γιούροβα. Με χαρά σας βλέπουμε εδώ την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Να μας θυμίζετε ότι η ισότητα δεν είναι απλώς αξία, αλλά και νομική υποχρέωση και θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Είναι και προς το συμφέρον μας. Είναι το μόνο που θα μας κάνει να προχωρήσουμε και να σκητρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες και να τις αφαιρώσουμε εκεί που πρέπει, δηλαδή να επιτύχουμε δυσότητα σε τούτο τον κόσμο. Αυτή η υποχρέωση δεν είναι απλώς βάρος για τις οικογένειες και για τις γυναίκες που θυμίζω ότι είναι και ε, πλειονότητα στον πληθυσμό αλλά ε, το 2016 βλέπουμε ε, να εξακολουθεί να ισχύει ένα τεράστιο μισθολογικό χάσμα κατά μέσο όρο 16% αλλά Στη χώρα μου αγγίζει το 25% την Ισπανία. Ε, η φτώχεια είναι περισσότερη για τις γυναίκες γιατί και στη συντάξη είναι τεράστιο το χάσμα. Και επίσης η οικονομική κρίση οδήγησε στο γεγονός ότι έχουν μικρότερη πρόσβαση και με χαμηλότερους μισθούς κάθε φορά οι γυναίκες. και παραμένει τεράστια ανισότητα στι ε, ηγετικέ και διοικητικέ σχέσεις των εταιριών. Για όλα αυτά υπάρχουν νομικά μέσα κυρίε και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και τονίζω το σύνεδο για να προχωρήσουμε σε αυτή τη νομική υποχρέωση που έχουμε να φτάσουμε στην ισότητα. Για το λόγο αυτό υπάρχει και η άδεια ε, μητρότητας, η, γονική άδεια, πατρική άδεια, όπως λέει, θέλετε πέστε το, αλλά εκκρεμεί μια ε, ευρωπαϊκή οδηγία, γι' αυτό και το οφείλουμε σήμερα στις οικογένειες. Θα πρέπει ε, να προχωρήσει και η οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες ε, μεταξύ αυτών είναι και η σημερινή Προεδρία που μπλοκάρουν. Το 40% δεν είναι καμιά ιδιοτροπία μας. Θα θέλουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την προσωπική σας δέσμευση κυρία Γιούροβα και σήμερα ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνυπογράψει και να ενταχθεί στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι το πρώτο βήμα για να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών. Ε, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Ε, η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την παρουσίαση ε, που κάνατε. Ε, όλες οι γυναίκες αγαπάμε τα λουλούδια, τουλάχιστον μερικέ, αλλά σήμερα δεν είναι μέρα για λουλούδια, είναι μια μέρα σήμερα για να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει για να πετύχουμε ε, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με έχει κουράσει λίγο αυτή η ετήσια εκδήλωση ενδιαφέροντος, γιατί είναι προφανές ότι η κατάσταση για τις γυναίκες, η κοινωνικονομική δεν βελτιώνεται στην Ευρώπη, η ανισότητα μεταξύ φύλων έχει αυξηθεί το ε, το, οι διαφορές ε, οι μισολογικές και ταξιδιωτικές αυξάνονται και 29 γυναίκες δολοφονήθηκαν στη χώρα μου ε, στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας πέρυσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισότητα η οποία δεν θα ξεπεραστεί με τα λόγια ή με ποσοστώσεις. Τώρα ήρθε η στιγμή να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά το θέμα και προφανώς αυτό που κάναμε μέχρι σήμερα απέτυχε και θα πρέπει να βάλουμε και τη γονική άδεια μητρότητας ή πατρότητας σε προτεραιότητα για να μην μείνουμε στα λόγια. Γιατί ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε πολύ άσχημα με ε, την άδεια μητρότητας και πατρότητας, ε, απορρίπτοντας τα κείμενα. Νομίζω ότι θα πρέπει τα λόγια που λέμε μια φορά το χρόνο να τα κάνουμε πράξη. Ράιντκε. Κύριε Ράιντκε. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Το 1959 γεννήθηκε η μάνα μου. Είχαν έξι παιδιά στην ε, οικογένεια και ζούσαν σε ένα ορεινό χωριό. Και κάτι άλλο έγινε. Πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Είχαμε τους ε, Έλληνες ηγέτες που κάπου στην Νότια Ευρώπη υπέγραψαν τη της Ρώμας. Σήμερα όμως δεν έχουν ακόμα κληρωθεί οι στόχοι αυτής της ε, συνθήκης γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ισότητα μηδής ανδρών και γυναικών την ίδια χρονιά γεννήθηκε η μάνα μου, αλλά και αυτή η αρχή της ισότητας. Παρ' όλα αυτά όμως ποτέ δεν απείλαψε αυτή την απόφαση, τους καρπούς αυτής της απόφασης η, μητέρα μου. Θα έπρεπε να αμυφθεί το ίδιο όπως οι άντρες για τη δουλειά που έκανε. Επομένως και σήμερα ακόμα υπάρχει ε, αυτό το χάσμα μεταξύ αμοιβών των δύο φίλων. Ε, ιδίω στη Γερμανία. Και έχουμε εκατομμύρια σκληρά εργαζόμενε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι οι εκείνες όπω και η μητέρα μου έχουν δικαίωμα να είναι αγανακτισμένε γιατί έχει αποτύχει 100% η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν μπορέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσουν αυτή την αρχή. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα και επομένω θα πρέπει να θυμηθούμε σήμερα ότι πρέπει να δώσουμε μάχη για την ισότητα τις ε, τελευταίες έξι δεκαετίες έχει προδώσει τις γυναίκες η Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε δεν θα πρέπει ε, εγώ και η γενιά μου που είναι πριν από 30 χρόνια να πιστεύουμε στην Ευρώπη αλλά να μην ε, έχουμε αυτό που μας αξίζει δηλαδή η ισότητα αμοιβή για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι σαφής η νομική βάση οπότε πρέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να προβούν σε τέτοια κίνηση οπότε δράσουμε τώρα και ας αυτή η αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πάρκερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Γύρω στα δύο ότι μεταξύ του 2010 και 2012 είχαμε 30.000 ανθρώπου που ήταν ε, δουλεμπορία και είχαμε 80% αυτών που ήταν γυναίκε και λένε επίση ότι και 3.000 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι είχαμε 21% αύξηση από την προηγούμενη χρονιά. Οπότε έχουμε αυτή τη καινούργια μορφή δουλειά και νομίζω ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μα έχετε ε, αναγκάσει να μην ε, έχουμε σύνορα οπότε αυτές οι συμμορίε δρούν ελεύθερα και λέει η κυβέρνησή μα ότι η ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλεύονται συνεχώ αυτέ οι συμμορίε και ασκούν αυτή τη δουλεμπορία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτέ οι κοινωνικέ πολιτικέ δυσκολεύουν την ε, ε, καταπολέμηση αυτών των ε, εγκλημάτων. Οπότε οι μόνοι που έχουν ωφεληθεί από όλε αυτέ τις κοινωνικέ πολιτικέ είναι αυτοί οι δουλέμποροι. Μπορείτε παρακαλώ να μιλήσετε πιο αργά γιατί είναι αδύνατον έτσι να μεταφραζείτε τους διερμηνείς. Λέει πρόεδρος. Πέστε μου, θέλετε να ξεκινήσω πάλι. Ρωτάει η κυρία Πάρκερ. Α, συνεχίστε τώρα. Κυρία Πάρκερ, συνεχίστε. Λοιπόν, οι μόνοι που ωφελήθηκαν ήταν οι δουλέμποροι και όλοι αυτοί που θέλουν να κακοποιούν και οι βία γιατί δεν μπορούμε να διερευνήσουμε το ποινικό τους μητρό όταν μπαίνουν στη χώρα. Εμείς ε, ανήκουμε στη Διεθνές εργασία Εργασίας και θέλουμε τις ε, ίσες συνθήκες εργασίας και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις υπηρεσίε του ΟΗΕ ε, για αυτόν τον σκοπό οπότε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους δεν θέλουμε να μην εφαρμοστεί η Άγια της Μητρότητας. Απλώς δεν θέλουμε οι κινδυνολόγοι να δικαιωθούν. Ε, αλλά όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα πετύχουμε που θέλουμε εάν αποχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Κάπελ, ευχαριστώ Πρόεδρε και οι γυναίκες ε, σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομία και την αμοιβή ε, υπολείπονται κατά πολύ. Διαφέρει η κατάσταση από κράτος σε κρότος ε, Παρ' όλα αυτά ισχύει. Παρόλο που οι γυναίκες ε, ε, είναι πάρα πολύ καταρτισμένες, σπουδαγμένες, μορφωμένες, δεν φτάνουν στις ηγετικέ θέσεις στις εταιρείας και έχουν αγωνιστεί και πάρα πολλά χρόνια για όλα αυτά. Κερδίζουν 16% λιγότερο από τους άνδρες. Η ψαλίδα αυτή σε κάποια κράτη-μέλη είναι μεγαλύτερη. 2,9% Σλοβενία, 6,5% στην Ιταλία, 22% ε, ε, στην Αυστρία, 28,3% στην Εστονία. Αυτό έχει μεγάλη σχέση με τα παιδιά, με τη μερική απασχόληση. Μία στι τρει γυναίκες που έχουν ε, παιδιά εργάζονται σε μερική απασχόληση. Ενώ στην Αυστρία την παρτίδα μου, ένα στους 20 άνδρες και όσο περισσότερα παιδιά έχει μια ε, μητέρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εργάζεται σε μερική απασχόληση. τα κέρδη ε, αυξάνονται, τα μερίσματα κατά 53% και τα κέρδη της εταιρείας κατά 42% σύμφωνα με μελέτες όταν υπάρχει γυναίκα σε διοικητικό συμβούλιο. Όσο περισσότερες είναι οι γυναίκες στην ηγεσία, τόσο αυξάνεται και ο τζίρος μέχρι 15%. Κατά μέσο όρο 5% όταν είναι στα υψηλά κλιμάκια γυναίκες. Αυτά είναι μελέτες από Ινστιτούτα σοβαρά. Ε, οι γυναίκες λοιπόν πραγματικά επιτέλους θα πρέπει να έχουν ίση εκπροσώπηση για αυτή που τους αξίζει και τους αναλογεί. Ευχαριστώ κυρία Μόρβαι. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα κι εγώ να πω ότι ε, είμαστε Στρασβούργο, 50 άτομα παρόντα από τους 700 τόσους βουλευτές, λες και είναι καμιά επέτειο σήμερα και καμιά πανηγυρική συνεδρίαση, η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Είναι ιδιαίτερη μέρα όμως, με ιδιαίτερα και ιστορική σημασία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να επιβάλλει ένα επέσχυντο σχέδιο και κατάπτυστο. Διότι παγκοσμίως βλέπουμε διάφορες βιοπραγίες, ε, ε, δεχθεί εγκλήματα κατά των γυναικών και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το χειραγωγήσει. Είναι πραγματικά επέσχυντη η ε, κατάσταση αυτή και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η μετανάστευση φέρνει πολλούς και γυναίκες στην Ευρώπη. Και τώρα έχουν καταλάβει οι θύνοντες και οι πολιτικοί και οι οικονομικοί ότι έχουν μπλέξει. Διότι ο κόσμος ε, στην Ευρώπη έχει κυριολεκτικά αγανακτήσει. Έχει μπουχτίσει και σου λέει δεν είναι κρίση προσφυγική, δεν είναι κρίση ασύλου, ούτε προσφυγικό είναι το θέμα, είναι μεταναστευτικό. Αυτά όμω όμως δεν είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσφυγική κρίση μπορεί να είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόλις το 10% των μεταναστών είναι πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από το ε, πόλεμο. Ποια είναι η λύση λοιπόν και τι βρήκανε. Θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Να δώσουμε ένα διαφορετικό καθεστώς στους πρόσφυγες. Εάν οι γυναίκες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και από τις διακρίσεις στη χώρα τους, γιατί αυτό είναι, τότε έχουν κάθε δικαίωμα να έρχονται στην Ευρώπη και να ζητούν άσυλο και αυτή τη στιγμή τους δοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και ε, μετά φέρουν και την οικογένειά τους για την επανένωση των οικογενειών. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα είναι η επόμενη φάση στην έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ που είναι παλιά μου φίλη και θα συζητήσουμε την έκθεσή της στη συνέχεια ότι οι πάντες έχουν ίδια ε, αξία ε, και τα πάντα είναι μια πρόφαση για να προωθηθεί αυτό το επέσχυντο σχέδιο. Στην έκθεση Χάνιμπολ το σημείο 13 είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ κυρία Βόζεμπερκ, παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά μιλάμε για την ανισότητα ή μάλλον για το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Δεν μας τιμά αυτή η συζήτηση, αλλά είναι ανάγκη να γίνεται. Σας τιμά, κυρία εκπρόσωπε, κυρία Επίτροπε, κυρία Γιούροβα, το γεγονός ότι υποστηρίζετε την οδηγία που αφορά στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πρόσφατα είχα την τιμή να παρουσιάσω μια έκθεση για τις γυάλινες οροφές, για το glass ceiling, τα εμπόδια δηλαδή που αρθώνονται στις γυναίκες αναφορικά με την επιδίωξή τους στα ανώτατα αξιώματα και τι παρατηρούμε οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται μόνο το 31% στην επιχειρηματικότητα ε, εκπροσωπείται από γυναίκες τις αυτοαπασχολούμενες ενώ ο στόχος όπως ξέρετε της στρατηγικής 2020 είναι να καλυφθεί περίπου το 75% αλλά η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι όπως προανέφερα σε όλα τα επίπεδα στις επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση στα ανώτατα αξιώματα στην επιστήμη την έρευνα την τεχνολογία τον ακαδημαϊκό κλάδο και πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο να αρθεί. δύο δρόμοι υπάρχουν το φυτόριο που λέγεται σχολείο το φυτόριο που λέγεται εκπαίδευση παιδεία το φυτόριο που λέγεται οικογένεια διότι αν οι προκαταλήψεις αυτές δεν αρθούν και αν δεν γεννηθούν καινούριε αντιλήψεις μέσα από την προβολή σωστών προτύπων και επιτευγμάτων των γυναικών τότε θα φτάσουμε πάλι σε πέντε χρόνια σε δέκα χρόνια να μιλάμε για ανισότητες. μια συζήτηση που διακρίνει τις γυναίκες από τους άντρες που δεν αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι και το μισό του πλανήτη είναι μια συζήτηση που δεν τιμά τις αξίες μας δεν τιμά τις αρχές μας δεν τιμά τη γυναίκα δεν τιμά την ευρώπη. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σε όλους. Στην ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κατοχυρωθεί η δέσμευση να επιτευχθεί ισότης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φέρει πολλά αποτελέσματα για να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Με νομοθεσία για την ίση αμοιβή, για τη γονική άδεια, για την άδεια για φροντίδα και προστασία για έγκυες εργαζόμενες, για να αναφέρω μόνο λίγα από τα άμεσα ωφέλη. Ξέρω ότι έγινε ε, δουλειά με αυτή την νομοθεσία και ε, χρησιμοποίησε ε, επί 20 χρόνια που ήμουν συνδικαλίστρια. Οι γυναίκες έχουν επωφεληθεί από αυτό και η χώρα μου με πληρωμές, με προστασία για τις γυναίκες και στις συντάξεις και στην εργασία. Ουδής όμως μπορεί να ισχυριστεί ότι επιτύχαμε τον αρχικό στόχο της ισότητας. Δεν μπορούμε και δεν ε, επιτρέπεται να επαναπαυόμαστε. Πρόσφατα είδαμε γυναίκες να υφίστανται ε, άνισα τις συνέπειες της λιτότητας και την απορρίθμιση της εργασίας που οδήγησε σε περισσότερες επισφαλείς εργασίες και μερικής απασχόλησης δουλειές. Βλέπουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 και υπάρχει συμφωνία βεβαίως ε, μεταξύ όλων ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ε, μείωση του μισθολογικού χάσματος και της ψαλίδας, ηγετικές σχέσεις για γυναίκες, εργασία γυναικών, μείωση της φτώχειας. Αλλά οι στόχοι στον τομέα αυτών χωρίς δράση δεν έχουν κανένα νόημα. Και αν κοιτάξουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι κατοποιητικά και αθαρρυντικά όλα αυτά δεν έχει γίνει πρόοδος ε, ούτε για την ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών, ε, ούτε για την οδηγία για τη γονική άδεια. Ωραία είναι αυτά που μας λέτε σήμερα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα σημερινά λόγια θα πρέπει να ακολουθούν από έργα όλες τις υπόλοιπες ημέρες του έτους. Ευχαριστώ η κυρία Χουισμένοβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όταν μιλάμε για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γυναικών θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη και το λόγο μεταξύ ε, παιδείας, ε, εισοδημάτων και δυνατοτήτων για ανέλεξη ε, στον επαγγελματικό κόσμο. Και παρόλο που είναι, ε, έχουν εξαιρετικά πολύ μόρφωση οι γυναίκες στην Ευρώπη, οι υπόλοιποι δείκτες υστερούν. Για να πετύχουμε λοιπόν μια βελτίωση χρειάζεται μια γρήγορη ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχουμε την ισότητα μέχρι το 2020. Σήμερα η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας είναι μια ευκαιρία για να θυμηθούμε πως πρέπει να στηριχθούν οι γυναίκες και η νέα στρατηγική θα πρέπει να, στρατηγική, να στηριχθεί από το Συμβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολιτικές που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη στοχευμένες έτσι ώστε η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γυναικών και η ισότητα μεταξύ ε, των φύλων να βελτιωθούν. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα με την αφορμή της Διεθνής της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτές τις ε, υποσχέσει μέσα από τι πολιτικές αλλά όμως η λιτότητα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα παρόξενε την ανισότητα οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν σε περισσότερη φτωχοποίηση και έχουν χτυπηθεί κατεξοχήν οι γυναίκε ανεργία, επισφαλής θέση εργασίας διακριτική μεταχείριση στο μισθολογικό αλλά βέβαια και σε σχέση με την άδεια ε, είδατε ότι αναγκάστηκε να κάνει πίσω Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το μέτωπο. Επομένω, θα πρέπει να πετύχουμε περισσότερη δικαιοσύνη, ισορροπία, περισσότερη ευελιξία. Να μην έχουμε αυτή την απορρίθμιση του χρόνου εργασία. Να μην δυναμητίζεται το κοινωνικό σύστημα και κοινωνικό πρότυπο. Έτσι θα πετύχουμε κοινωνική ε, πρόοδο, αλλά και κυρίω χωρί πολιτική λιτότητα. Κύριε Αγίουτο, ευχαριστώ, Πρόεδρε θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό συνάδελφοι για το πώς έχει η κατάσταση των γυναικών γιατί αν το κάνουμε θα διαπιστώσουμε ότι προχωράμε σημειωτών γιατί βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί στη με των γυναικών. Δεν υπάρχουν δυνατότητες πραγματικής, αυθεντικής επιλογής για τις γυναίκες. Άρα θα πρέπει η γυναίκα να έχει την ελευθερία της επιλογής, να διαλέξει να σπουδάσει όπου θέλει, να μπορεί να διαλέξει ένα, ένα επάγγελμα, αλλά να μην κυριαρχούν οι άντρε Γι' αυτό γίνεται και στι επιχειρήσεις και στην πληροφορική. Να μπορέσει όταν θέλει να κάνει παιδί. Όμω όμως ε, σπρώχνονται στην ανεργία και θα πρέπει ο η πολιτική να δώσει κάποια απάντηση για αυτό το έτοιμο των γυναικών και βλέπουμε ότι απέτυχε αυτή η οδηγία απέτυχε η θέσπιση της οδηγίας για το, την άδεια μητρότητος επομένως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει ε, μια σταδιοδρομία και αυτό να μπορούν να το έχουν και οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι ε, να καλυφθούν και να τους φροντίσουν. Οι γυναίκες επομένως θα πρέπει θετικά να προσπαθήσουμε να υπάρξουν ελπίδες στο μέλλον, η Πρόεδρος. Και τώρα και Σκορδίνη Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, οι επιστήμονες έχουν μελετήσει ε, τους Αμερικάνους μπασκετβολίστες και ε, είπαν ότι είναι καλύτερα να είσαι ψηλό για να παίζει μπάσκετ παρά να είσαι κοντός. Ε, λοιπόν, όταν πληρώνονται οι γυναίκες ε, λιγότερο ή φτάνουν σε χαμηλότερες θέσεις από τους άνδρες στις εταιρείες σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά ικανές ή δεν έχουν την ευκαιρία. Οι γυναίκες είχαν την ευτυχία να μεγαλώνουν τα παιδιά τους που ήταν ευλογία και ξαφνικά αποφάσισε κάποιο ότι οι γυναίκε πρέπει να εργάζονται και τα παιδιά να πηγαίνουν σε βρεφονιπιακού σταθμού και σε παιδικού πριν το σχολείο και έχουν πέσει οι αποδόσει παντού. Θα πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται στο bridge, στο σκάκι ε, και στα άλλα αθλήματα υψηλού επίπεδου. Οι γυναίκε είναι μόλι το 1%. Και μήπως όλη αυτή η πίεση είναι τεχνητή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι φυσική ε, έχει πέσει και το επίπεδο των παιχνιδιών και εκτός από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστραφεί. Ε, ε, έχετε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Γιάκοψη. Θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής κύριε Κόρβεν Μίκε. Πρέπει να σας πω ότι έπαιζα εξαιρετικό μπάσκετ και όπως βλέπετε δεν είμαι και πάρα πολύ ψηλός. Ε, αλλά πραγματικά έπαιζα εξαιρετικό μπάσκετ. Το ξέρετε αυτό εσείς και ξέρετε τι χρειάζεται. Το αποφασιστικό δεν είναι το ύψος, είναι η τεχνική. Είναι αν μπορείς να βάζεις καλάθια ή όχι. Και το ίδιο ισχύει για όλα τα υπόλοιπα που είπατε. Συμφωνείτε ότι δεν είναι ε, στο μπάσκετ αποφασιστικό το ύψο. Μία μόνο μπλε κάρτα, είναι πάρα πολλέ. Συνεχίζουμε, λέει η Πρόεδρο. Α, ναι, ναι, πρέπει να απαντήσετε, βεβαίως, προφανώς. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πληροφορήσω πως οι υψηλοί άνδρες δεν κερδίζουν περισσότερο από τους κοντούς. Άρα λοιπόν είναι άδικο αυτό. Και εγώ έπαιζα ε, στην Πολωνία μπάσκετ και πρέπει να σας πω πως ήμουν στη Β' Εθνική και την πρώτη Εθνική Γυναικών την κερδίζαμε με 50 πόντους διαφορά. Τέρα. Grazie Presidente. L'8 marzo ci ricorda ogni anno quanto ancora deve essere fatto per migliorare... Τις 8 Μαρτίου πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα πρέπει να κατάσταση για τις ε, Ευρωπαϊκές υπάρχουν πάρα πολλοί βραγμοί ούτω ώστε να υπάρχει ισότητα για τι γυναίκε στην κοινωνία μα και εμεί, ω νομοθέτε, επιβάλλεται να μπορέσουμε να ε, πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Πρέπει για να φτάσουν την αμοιβή των μισθών θα έπρεπε να δουλεύουν δύο μήνες παραπάνω οι γυναίκες επομένως υπάρχει ανισορροπία αλλά υπάρχει και στις ε, συντάξεις και αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες γυναικών ε, κινδυνεύουν να πέσουν σε φτώχεια Επίσης υπάρχει μεγάλη απειλή φτώχειας ε, για τις ηλικιωμένες, πολύ περισσότερο από για τους ηλικιωμένους. επομένω θα πρέπει να αρθεί αυτή η ανισότητα και ε, προσπαθούμε να το αποτύχουμε αυτό και στην ε, Επιτροπή Θεμάτων Γυναικών και Ισότητας. Οπότε είδαμε ότι αυτή η έκθεση την οποία κατέβασα συγκέντρωσε πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία ακριβώς για να δούμε ε, πώς θα μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετάσχουν περισσότερο στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη αλλά είπαμε ότι θα... μιλάμε για το 1 τρίτον των γυναικών που να, είναι επιχειρηματίες όμως ε, είδαμε ότι οι γυναίκες που έχουν ε, πληγεί είναι 63% από το 60% που ήταν πριν οπότε θα πρέπει να πούμε μπράβο στην Επίτροπο κυρία Γιρόβα για τις προσπάθειές της. Οπότε θα πρέπει η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης να προσπαθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Έχετε μια επερώτηση. Δέχεστε μάλιστα. Κύριε Τσάντζη. Ε, Κύριε Τζένι σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ερωτήσω το εξής. Ας κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομία αν επιτρέπετε. Διότι 8 Τρίτου είναι η Παγκοσμία Γυναίκας το 1917 του χρόνου επομένως θα είναι η εκατοστή παγκοσμία της γυναίκας που θα ερωτάζουμε. Οπότε φυσικά και πρέπει να υπάρχει ισότητα μισθολογική αλλά προστασία γυναικών και ανηλίκων. Αλλά και ένας άλλος στόχος είναι η παρουσία συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνία του χρόνου θα πρέπει σαν ε, τέταρτο στόχο να έχουμε την ε, πάυση και τα πολέμηση τη βία και των γυναικών. Συμφωνείτε κύριε Ματέρα που έχει το λόγο. Νόμιζα ότι πρόκειται για ερώτηση. Αλλά τελικά ήταν ε, παρατήρηση, παρέμβαση του συναδέλφου. Δεν καταλαβαίνω τι ρωτήσατε. Όλα αυτά σας άκουσα. κάθε μέρα με ένα τέτοιο αγώνα, ώστε όλε οι χώρε να ακυρώσουν την, τη σύμβαση του Κωνσταντινούπολη, ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο τη βία κατά γυναικών και ανηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Και σα ευχαριστώ. Πρόεδρο. Η κυρία Πόστη είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς δεν σεβόμαστε με τον και τρόπο την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκε δεν κερδίζουν τα ίδια χρήματα με του άντρε, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην αγορά εργασία, δουλεύουν πιο πολύ, έχουν ε, πολύ περισσότερου όρου εργασία που δεν πληρώνονται, είναι πιο φτωχέ. Και οι ηλικιωμένε γυναίκε αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ δυσκολίε και δεν έχουν καταφέρει να απολαύσουν τα δικαιώματά του στο παρελθόν. Άρα λοιπόν έχουμε διακρίσει. Μία γυναίκα Ρώμα αντιμετωπίζει διακρίσεις γιατί είναι γυναίκα αλλά γιατί έχει και προβλήματα ρατσισμού. Μία γυναίκα, η ΛΟΑΔ, ε, αντιμετωπίζει διπλή δια, διακρίσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει όταν συζητάμε για τέτοιου είδους πολιτικές να διαπιστώνουμε πως το όλο σύστημα είναι άδικο, πως υπάρχει κόστος και ανθρώπινο και οικονομικό από αυτές τις διακρίσεις και υπάρχει μια συνεχιζόμενη καταπάτηση δικαιωμάτων η οποία γίνεται αποδεκτή από εμά και για την οποία δεν κάνουμε τίποτα εδώ και καιρό. Βλέπω πως για σας η πολιτική αυτή δεν είναι προτεραιότητα. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως η ισότητα είναι ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα, ενώ θα έπρεπε να έχουμε μια πιο καλά πλαισιωμένη στρατηγική έτσι ώστε οι γυναίκες και οι άντρες ε, στην Ευρώπη να μπορούν να αποφασίζουν με τον ίδιο τρόπο για τη ζωή τους. Είμαι φεμινίστρια και το θεωρώ παράδεκτο. Θα πρέπει η ισότητα να αποτελέσει μια απόλυτη προτεραιότητα. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για εμάς. Πώς θα ήταν ο κόσμος εάν το μισό του πλανήτη μας εξακολουθεί να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να το ξεπεράσουμε και προσωπικά να σας πω πως εγώ δεν γιορτάζω στις 8 Μαρτίου γιατί θεωρώ πως η γιορτή αυτή αποτελεί απλώς λόγια ε, που υπογραμμίζουν τις ανισότητες που ακόμα ισχύουν και αποδεικνύει πως 364 από 365 ε, μέρες το χρόνο δεν γιορτάζουν οι γυναίκες. Η κυρία Χέντε σας έχει ζητήσει ε, μπλε κάρτα. Ε, κυρία μου, τη δέχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα απόλυτα με τα όσα είπε η Σοράγια Πόστ και εγώ δεν γιορτάζω την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Γιατί? Γιατί θεωρώ πως θα έπρεπε να είναι η Μέρα της Γυναίκας κάθε μέρα και πως θα έπρεπε να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να το πετύχουμε. Πείτε μου, συνάδελφε, θεωρείτε πως υπάρχει κάποια στρατηγική, σαν αυτή που είχε στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να πετύχουμε την ισότητα αυτή. Πιστεύετε πως χρειάζεται μια στρατηγική ε, που θα εφαρμοζόταν για όλους, θα ήταν πιο αποτελεσματική από ένα απλό έγγραφο. Ναι, ε, είμαι σίγουρη. Νομίζω πως θα πρέπει να στείλουμε ένα πολύ στεναρό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη. Πιστεύω πως η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει ε, να αποτελέσει προτεραιότητα και να μην έχουμε απλά ένα έγγραφο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και άλλη μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Ε, κύριε Βάουτμαν, θα πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, ε, ε, το μικρό μου φρόνο δυστυχώς δεν λειτουργεί, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε λίγο πιο πικάντικη τη συζήτηση. Τι είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, χρειάζεται. Ακόμα δύο συνάδελφοι είπαν ότι δεν χρειάζεται και αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Ακούσαμε από την Επίτροπο ότι ως γυναίκες θα πρέπει να εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για ίσα δικαιώματα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Κάθε μέρα κανονικά, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Αλλά ας παρακαλώ θα πρέπει να αναδεικνύουμε τον αγώνα αυτό τη σημερινή ημέρα. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει και η ε, άδεια εγκυμοσύνη, η μητρική άδεια να γίνει γονική άδεια για να μπορούν οι γυναίκες να αναπτύσσουν και τη σταδιοδρομία τους με την άνεσή του και με τον τρόπο που θέλουν. Απάντηση. Βε, βεβαίως, ε, συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε θα πρέπει να ε, υπάρχει όχι άδεια εγκυμοσύνης αλλά γονική άδεια που να μοιράζονται ακριβώς ε, οι ε, άνδρες με τις γυναίκες. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη σχέση γι' αυτό με την 8η Μαρτίου. Θα πρέπει καθημερινά και 24 ώρες το 24ωρο να αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία στην οποία θέλουμε να τρέφουμε τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, με τον ίδιο τρόπο να αξιοποιούν όλοι το δυναμικό τους και τις ικανότητές τους ε, από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής τους. κυρία Κοζάλες. Ευχαριστώ πολύ. Το να, καταπολεμήσουμε αυτή την ανισότητα στην Ευρώπη είναι μια μάχη που χρειάζεται να δίδεται κάθε μέρα και όχι μόνο στις 8 Μαρτίου. Υπάρχουν τρία στοιχεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Πρώτα απ' όλα η ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελλειπή παρουσία των γυναικών στα κέντρα εξουσίας. Στο Κοινοβούλιο για παράδειγμα, 10 από τις 25 επιτροπές έχουν πρόεδρο γυναίκα. Δεύτερον, εμείς έχουμε υποστεί τις χειρότερες εργασιακές συνθήκες έχουμε ποσοστά ανεργίας υψηλότερα, μεγάλες διαφορές και, στα, και στις ε, μισθούς και στις συντάξεις πάνω από το 16% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αναλαμβάνουμε το βάρος της φροντίδας. Μία αόρατη δουλειά που είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός. Και τέλος, οι διαφορές οξύνονται μεταξύ βορρά και νότου στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε τις πολιτικές λιτότητας που επιβαρύνουν διπλά τις γυναίκες. Η χειροτέρευση των δημοσίων ε, ε, δομών πρόνοιας οδηγούν στο να αντιμετωπίζουμε εμείς τα χειρότερα φαινόμενα που προκαλεί η λιτότητα. Η Ευρώπη ζητά ισότητα και εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημά της αυτό. Η κυρία Κραπίνη έχει μία μπλε κάρτα για εσάς. Μπορείτε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σας άκουσα να μιλάτε και εσάς και άλλους συναδέλφους για την ανισότητα αυτή και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα είναι, η πλειονότητα του πληθυσμού είναι γυναίκες. Γιατί δεν ψηφίζουν οι γυναίκες άλλες γυναίκες. Το πρόβλημα είναι ότι ε, στην εξουσία δεν την έχουν οι γυναίκες. Ε, ε, πλειονότητα εκείνων που ασκούν εξουσία είναι άνδρες. Για να μην πω ότι η ανισότητα και η ε, ανδροκρατία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα κοινωνιολογικά. Θα πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα και με συγκεκριμένα χρήματα και πόρους. Ευχαριστώ, η κυρία Σόιντροπα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσουμε την κυρία Επίτροπο διότι η προσέγγιση της είναι πάρα πολύ επιτυχημένη και πάρα πολύ σωστές οι συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε για την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Είδαμε τι έχει γίνει με αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Είδαμε ότι η κατάσταση των γυναικών δεν είναι καθόλου αυτή που θα θέλαμε. Και στην ε, Τσεχία υπάρχει ε, μισθολογικό χάσμα πάνω από 12% και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ο λόγος ποιος είναι. Οι γυναίκες κάνουν δουλειές που γενικά αμείβονται λιγότερο όπως δασκάλες ή νοσοκόμες αλλά επίσης οι γυναίκες φροντίζουν τα παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας που χρειάζονται περιποίηση και βοήθεια. Ε, τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τις ε, γυναίκες, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε και τις γυναίκες οι οποίες γίνουν ένα ή και περισσότερα παιδιά, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί γενναιότητα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη οικονομική πλαισίωση, οικονομική ασφάλεια εκτός από την άδεια. Οπότε θα πρέπει να αποδείξουμε με αυτόν τον ε, σεβασμό μας ότι δηλαδή και μετά τη γεννησία παιδιού να μπορεί η γυναίκα να δράσει στην αγορά εργασίας ε, να είναι προστατευμένη από βλαπτικές ενέργειες κάποιου εργοδότη. Να μπορεί η γυναίκα να έχει δουλειά. Ευχαριστώ προς τη μάνα μου γιατί ξέρετε ήταν ε, η τέλεια μητέρα αλλά και η ιατρός. Έχετε μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Από τον κύριο Φουντούλη. Θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ κύριε Φουντούλη. Ευχαριστώ. Οι απαιτήσει τη σημερινή καταναλωτική κοινωνία έχουν οδηγήσει τις γυναίκε σε έναν αγώνα δρόμου για επαγγελματική καταξίωση. Όμω οι γυναίκε έχουν το θείο δώρο του να γεννούν παιδιά η τωρινή οικονομική κατάσταση του επιτρέπει να κάνουν το πολύ ένα παιδί. έτσι λέμε ότι η ευρώπη γερνάει. δεν θα έπρεπε να στηριχθούν οι οικογένειες οικονομικά έτσι ώστε οι μητέρες να μπορούν να ασχοληθούν οι ίδιες με τα παιδιά τους; έχουν ερωτηθεί; υπάρχουν στοιχεία για το τι θέλουν οι περισσότερες γυναίκες; μήπως αυτά που συζητάμε είναι αυτά που θέλουν οι γυναίκες καριερίστες; ευχαριστώ κυρία Σόντροβα. αξιότιμη συνάδελφε, Νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες θα πρέπει να είναι ε, σε θέση να αξιοποιούν το δυναμικό τους. Όταν λέμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι, είναι εξίσου ελεύθεροι και θα πρέπει να έχουν ευκαιρία να επιλέγουν ελεύθερα. Και βέβαια εγώ κατανοώ ότι οι γυναίκες είναι μητέρες και ε, να επιλέγουν οι ίδιες όμως να έχουν παιδιά και να μένουν σπίτι αν θέλουν, αλλά αν επιθυμούν να ε, κάνουν παιδιά και να επιστρέφουν στην καριέρα τους. Απουσιάζει η κυρία Πιτσέρνο. Όχι. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την Επίτροπο για την προσπάθειά της, αλλά και όλες τους συναδέλφους και τους συναδέλφους που θέλουν να συμμετάξουν σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το ότι σήμερα ε, δεν είναι κάτι το συνδυσμένο ε, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό επομένως καθημερινό για τις γυναίκες όλες γιατί οι γυναίκες είναι το μέλλον της Ευρώπης και εννοώ τις γυναίκες πρόσφυγες. Μιλάμε για 60% των προσφύγων που αποτελούν αυτή τη ροή των προσφύγων που περνάνε τα ελληνικά και μακεδονικά σύνορα. Οπότε τι νόημα έχει να εορτάζουμε κάτι για το παρελθόν ενώ τους κλείνουμε την πόρτα στο μέλλον. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα ωφεληθούν οι γυναίκες, πώς ε, θα σταματήσουμε να αγνοούμε ε, αυτού του είδους την ε, διακίνηση, την δουλεία που υφίστανται. Είναι ντροπή, είναι βία αυτό που περνάνε, άρα θα πρέπει η σημερινή επέτειος να κρυφθεί σε εκείνε, σε αυτές που φεύγουν, που είναι πρόσφυγες, που αναζητάνε μια ελευθερία που σήμερα θα πρέπει να θυμηθούμε. Εμεί πιστεύουμε σε μια διαφορετική αλληλέγγυα Ευρώπη και για αυτό το λόγο ε, θέλουμε να κάνουμε για άλλη μια φορά το ίδιο, δηλαδή μια επιστολή προς όλους. Να κάτσουμε να δούμε πώς ε, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση, καταπίεση, βία όλες αυτές οι γυναίκε που συνοθούνται στα μακεδονικά σύνορα. Τα βλέπουμε αυτά, τα έχουμε δει με τα μάτια μας, θα πρέπει να πάμε και να δούμε πώ υλοποιείται αυτό το όχι που λέει ο Ευρώπη, πρόκειται για ένα λάθο που είναι ένα τρόμος. Έχετε μια επερώτηση, θέλετε να απαντήσετε από τον κύριο Έθεριτζα. Κυρία Έθριτζ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσετε μαζί μου πως όλες αυτές οι τεχνητές εορτές όπως οι Παγκόσμιοι Μέρες της Γυναίκας δεν έχουν καμία σημασία και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν ευκαιρίες για όλους και να μπορούν οι γυναίκες στο δυτικό κόσμο να απολαμβάνουν τις δυτικές ελευθερίες και όχι αυτές να εξαφανιστούν με την πλημμύρα των ε, νέων λαών που καταφθάνουν στην Ήπειρό μας που έχουν διαφορετικές αξίες. Άρα λοιπόν οι, οι ευκαιρίες και η, δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες στη Δύση να ζήσουν όπως επιθυμούν να μην ε, από την είσοδο αυτών των νέων πληθυσμών στην Ευρώπη. Μπορείτε να απαντήσετε. Δεν συμφωνώ με τίποτα από όσα είπε και από τις λέξεις που χρησιμοποιήσει ο συνάδελφος γιατί πρόκειται η αυτή την παγκόσμια ημέρα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι κάτι ε, αυτή η επέτειο που μας οδηγεί να τιμούμε τις κατακτήσεις. Το τι κατάφεραν οι γυναίκες πριν από εμά που έδωσαν τον αγώνα τους ούτω ώστε εμεί να μπορούμε να απολαύσουμε τα αποτελέσματα και που θα πρέπει να θυμόμαστε το δικαίωμα στην ψήφο, το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στην μητρότητα. Είναι όλα αυτά τα οποία καμιά φορά τα θεωρούμε σήμερα αυτονόητα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ε, λέμε μεγάλες ε, κουβέντες για τις ελευθερίες δηλαδή Όμως η ε, υποχρεωσή μας να θυμόμαστε ότι αυτή η μεγάλη Ευρώπη την οποία εορτάζουμε και τιμούμε στην Κυριά Ήπειρο ήταν στο παρελθόν ένας φάρος αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν κάνει το καθήκοντας κλείνουμε τα μάτια σε όλα αυτά τα φρικτά σε αυτές τις ε, σκηνές που γίνονται, που λέμε για παιδιά, για γυναίκες που έχουν συνοδηθεί εκεί μπροστά σε ένα σειρματόπλεγμα και δεν μπορούν να έχουν τη ζωή που τους αξίζει, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε αυτή τη μέρα μνήμης, αλλά, αλλά θα πρέπει τόσο από αυτήν να έχουμε και μία μέρα ντροπή για όλους μας και διακόπτει το μικρόφωνο η Πρόεδρος. Sorry, but Συμπαθάτε με λέει η πρόεδρος, αλλά έχετε μόνο μισό λεπτό για να απαντήσετε. Και το, το υπερεύετε. Τώρα, διαδικασία κάτσε διάρε. Κύριε Μαριάννα Πέτυρ έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι οι γυναίκες είναι σε πολύ δινή θέση όταν ε, ζητούν δουλειά δεν τους υποστηρίζει κανείς για να τους βοηθήσει να ε, συμφιλειώσουν ε, την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Όταν χάνουν τη δουλειά τους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και όταν έχουν δουλειά ε, αμείβονται λιγότερο για την ίδια δουλειά από τους άνδρες. Υφίστανται παρενοχλήσεις και αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα. Παρόλο που οι πτυχιούχοι είναι γυναίκες στην πλειοψηφία τους στη συνέχεια δεν τις ξαναβρίσκουμε τις γυναίκες αυτές ε, στις θέσεις αποφάσεων. Πολύ συχνά δεν έχουν ε, σύνταξη, δεν έχουν περιουσία κίνητη και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Χρειάζονται τέτοια συνταξιδοτικά συστήματα που να προλαμβάνουν την φτώχεια των γυναικών. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ κυρία πρόεδρε εν ώψη του σημερινού εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης που διανύουμε και κυρίως στις χώρες που έχουν φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια οι γυναίκες είναι τα μεγαλύτερα θύματα καθώς τα δικαιώματά τους θίγονται καθημερινά τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο. συγκεκριμένα στον εργασιακό χώρο διαπιστώνεται ένα μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα που ανέρχεται στο 16,4% και ένα αντίστοιχο συνταξιοδοτικό χάσμα που ανέρχεται στο. 39%. Επιπλέον στους χώρους εργασίας παρατηρούνται διακρίσεις όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα που πλήττεται από τα μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητας, το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο έχει οθήσει τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες να διαθέτουν πάνω από το 80% του ετήσιου εισοδήματός τους για κοινωνικές για εισφορές και φόρους, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και οι αγρότησε προκειμένου η ευρωπαϊκή ένωση να θέσει τέλο στι διακρίσει που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλλα θα πρέπει να σταματήσει να φτωχοποιεί τι χώρε του ευρωπαϊκού νότου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μια ε, ουσιαστική πολιτική ισότητας για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα αίτια της κρίσης που μπορεί να είναι οικονομικά αλλά και πολιτιστικά. Να σας μιλήσω λίγο για αυτό το στοιχείο της νοοτροπίας και της κουλτούρας. Υπάρχει ε, διάκριση θεσμοθετημένη σε κάποιους χώρους όπως είναι η Καθολική Εκκλησία που εξακολουθεί να μην χειροτονεί γυναίκες. Ε, απλώς επειδή είναι γυναίκες. Αυτό δεν είναι διάκριση με βάση το φύλλο. Η Καθολική Εκκλησία ε, έχει οργάνωση τύπου κράτους και έχει και κράτος ολόκληρο τον Πατικανό ε, και θα πρέπει να παρακαλέσουμε τον ε, Ποντίφικα που είναι και αρχηγός κράτους να τερματίσει αυτή την αφόρητη διάκριση εις βάρος των γυναικών αν γίνει κάτι τέτοιο θα αποτελέσει τεράστια πρόοδο. Τουλάχιστον ε, για να μην έχουμε τέτοιες διακρίσεις με βάση το φύλλο. Κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο. κύρια Πρόεδρε, θα προτιμούσα πριν από μένα να λάβει το λόγο ο κύριο Στετίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να σα πω πω εκ μέρου των ανδρών δηλώνω πω ο σοβινισμό δεν αποτελεί κομμάτι του αυτού όλων μα. Και αυτό που ακούσαμε από διάφορου συναδέλφου με, με λύπησε και θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλε τι γυναίκε για την ημέρα τη γυναίκα. Και να προσθέσω πω 52% τη κοινωνία μα είναι γυναίκες. 48% είναι οι άνδρες. Η φύση αποφάσισε. Και παρόλα αυτά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συνέχεια διακρίσεις στην αγορά εργασίες, στις συντάξεις, στους μισθούς. Αυτό είναι η πραγματικότητα και πρέπει κάτι να κάνουμε. Και χαίρομαι που συνεχίζει το διάλογος για τα θέματα αυτά. Η Επίτροπος κυρία Γιούροβα πολύ συχνά συμμετέχει στις συζητήσεις αυτές. Παρόλα αυτά θα ήταν καλό ό,τι λέμε σήμερα εδώ στην αίθουσα να είναι αντιπροσωπευτικό ε, της κατανόησης που έχουμε για τη θέση της γυναίκας. Και δυστυχώς τα λόγια κάποιων συναδέλφων δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως οι άντρες χαίρονται που σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας και χαίρομαι που έχω σήμερα την ευκαιρία να πω δύο λόγια για το θέμα. Είναι σημαντικό να γίνει μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη οργάνωση ή θεσμός παγκοσμίω που να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών και γι' αυτό γίνεται και η συζήτηση εδώ άλλωστε. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε ε, μέχρι σήμερα αλλά ακόμα πρέπει να κάνουμε πολλά. Στη δική μου χώρα έγινε Έγιναν εκλογέ την περασμένη εβδομάδα και το 30% των ε, γυναικών που είχαμε στις, ε, στα ψηφοδέλτια μας μας οδήγησαν στο να έχουμε ένα κοινοβούλιο με μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών από ό,τι ποτέ. Άκουσα χτες δε στο ραδιόφωνο πως πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν περισσότερες γυναίκες στα συμβούλια τους με μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό είναι ένα δίδαγμα για όλους μας. Ναι. Ε, κυρία Γκέισνερ, ευχαριστώ ο Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι καταρχάς που βλέπω τόσους άνδρες εγώ εδώ γιατί ε, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους η ανισότητα. Σήμερα μιλούμε για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αλλά θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Δεν είναι επέτειος πανηγυρική για γιορτή η Παγκοσμία Μέρα της Γυναίκας, αλλά για απαιτήσει και διεκδικήσεις. Ε, πριν από 40 χρόνια αποφασίσαμε να υπάρχει ίση αμοιβή για εργασία και παραμένει η ψαλίδα 16%. Στη Γερμανία 22% και είναι η ντροπή μας αυτό. Και να μην μιλήσω για τις συντάξεις που είναι 39% και ε, είναι παράδεκτα πράγματα όπως και η βία κατά των γυναικών. Οι, οι γυναίκες είναι και αυτοί οι άνθρωποι όπως και οι άνδρες και δεν θα πρέπει να προστατεύονται. Και πρόσφατα μιλήσαμε και για την επιχειρηματικότητα των γυναικών και είδαμε ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ε, ενώ οι άνδρες είναι πιο εύκολο να δανειοδοτούνται έχετε την πλήρη μας υποστήριξη κυρία Επίτροπε. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική καινούρια που να είναι πραγματικά χρήσιμη και ωφέλιμη. Ο κύριος Καπούτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα 8 Μαρτίου είναι πάρα πολύ αυτό να συζητούμε για την κοινωνική κατάσταση των υγειών στην Ευρώπη. Παρ' έχουμε αυτέ τι δύο ε, οδηγίε που ε, αφορά τι ε, ευκαιρίε των γυναικών και δεν κατάφεραν να άρουν αυτό το κενό και να φέρουν την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων γιατί οι γυναίκε και στην Ευρώπη υφίστανται ανισότητα κοινωνικονομική άρα χρειάζεται να γίνει διόρθωση πορείας και να υπάρχει μια στρατηγική αυτό που ξέρει το 2015 είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και την γυναική ταυτότητα γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, παρουσία των γεγονών στα κέντρα και στα όργανα αποφάσεων. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις ε, ε, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και στην πολιτική. Θα πρέπει να έχουν το χώρο τους οι γυναίκες. Θα πρέπει να σταματήσουμε να περιζόμαστε στην Ευρώπη σε απλές καταγγελίες. Θα πρέπει να εμποδίσουμε τις δεμινές διακρίσεις βάρος των γυναικών και ελπίζουμε ότι στις επόμενες χρονιές θα γιορτάσουμε την 8η Μαρτίου και θα έχουμε λιγότερο χάσμα που θα πρέπει να γεφυρώσουμε. Ευχαριστούμε. τίνα. Ευχαριστώ. Ξέρετε, στάθηκα τυχερός στη ζωή μου γιατί συνάντησα πολλές ισχυρές, αποφασιστικές γυναίκες μεταξύ των οποίων ήταν και η μητέρα μου. Και ξέρετε, στον πόλεμο αυτοί που πέφεραν περισσότερο ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω σήμερα. Την ε, Παρασκευή που πέρασε η Νάντια Σεφτσέγκο απήχθη. Είχαμε και απεργία πείνας και σήμερα που έχουν περάσει πέντε μέρες συνεχίζει αυτή την ε, απεργία της δεν ε, πίνει επομένως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αυτό γίνεται γιατί πρόκειται για κάποια άδικη δίκη στην οποία έχει παραπενθεί. υπάρχει αυτή η ποινή βάση των 33 ετών, οπότε παρακαλώ κάντε ό,τι μπορείτε τόσο ώστε να απελευθερωθεί αυτή η γυναίκα. Κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα χαίρομαι πάρα πολύ και εκτιμώ κάθε ευκαιρία που έχουμε να συζητούμε στο Κοινοβούλιο τέτοια θέματα φύλου και πολιτικής ε, φύλου γιατί είναι σημαντική έμπνευση πάντα για τις εργασίες μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, σε σχέση με τα όσα είπατε, να σας απαντήσω. Ε, σε ό,τι αφορά την συμφιλίωση του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο, είπατε για την οδηγία για την γονική άδεια. Την αναθεωρήσαμε για να καταθέσουμε μια καλύτερη πρόταση που να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των γονέων. Διότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί η κατάσταση με την ε, οδηγία για τη μητρική ε, άδεια, γιατί τα κράτη-μέλη μας έλεγαν ότι αυτά ισχύουν ήδη στην νομοθεσία μας. Χρειαζόμαστε κάτι καινούριο, κάτι πιο σύγχρονο. Και γι' αυτό προετοιμάζουμε το πακέτο αυτό για το 2016, το νομοθετικό. Θα έχουμε μία δέσμη προτάσεων νομοθετικών και μη που θα βελτιώσουν ε, την ε, ζωή και των δύο γονέων. Εκτός από τα όσα είπατε εδώ, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι γυναίκες και να μην τους επιβάλλει κανείς, να μην τους υπαγορεύει κανείς τίποτα ούτε ε, υποτιμά, δεν είναι η πρόθεσή μας να υποτιμήσουμε το ρόλο των μητέρων, αλλά πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Πολλές νέες γυναίκες που έχουν βγάλει πανεπιστήμιο και είναι 60% οι πτυχιούχοι οι γυναίκες, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα κάνουν καριέρα ή οικογένεια. Οι παιδιά, έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Και από πλευράς οικονομικής ε, αυτό είναι παράλογο θα πρέπει να δημιουργούμε εμεί εκείνες τι προποθέσει που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να κάνουν και παιδιά και καριέρα. Και μάλιστα με υψηλά προσόντα και δεξιότητες. Δεν μας αρέσει αυτό που λέτε ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας να κάνει παιδιά και βέβαια είναι. Και εγώ μητέρα είμαι. Και ο πρώτος μου ρόλος στη ζωή μου ε, και ο βασικότερος είναι αυτός, της μητέρας. Παρ' όλα αυτά ζούμε σε μια κοινωνία η οποία βεβαίω χρειάζεται παιδιά, για να το πω με όρου πάρα πολύ κοινικού και οικονομικού. η κοινωνία χρειάζεται και παιδιά και χρειάζεται μελλοντικού φορολογούμενους. Γι' αυτό χρειάζεται παιδιά. Αλλά γιατί να ε, αναλαμβάνουν αυτό το φορτίο και από το βάρο μόνο οι γυναίκε. Αυτά δεν είναι επιλέον βιώσιμα πράγματα. Γι' αυτό προσπαθούμε να ε, εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή για τη νέα δέσμη για να έχουμε και νέα στοιχεία, όχι μόνο καλύτερες ε, διευθετήσεις για τις γυναίκες, αλλά για τους εργαζομένους γονείς. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι το αποτέλεσμα των προτάσεών μας. Βεβαίω υπάρχει μισολογική ψαλίδα και χάσμα και θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέσα για να μειωθεί αυτή, να κλείσει. Έχετε δίκιο. Κατά μέσο όρο είναι 16% η διαφορά στι αμοιβέ. Είναι πολύ ψηλή και σε ορισμένα κράτη-μέλη ακόμα υψηλότερη. Είπαμε το 16% είναι μέσο όρο. 39 και 40% ε, ψαλίδα της συντάξεις. Αυτά τα πράγματα είναι αφόρητα πλέον. Και εγώ εξακολουθώ να πιέζω τα κράτη-μέλη να εντάξουν στην κοινωνική τους και φορολογική τους νομοθεσία εκείνα τα μέτρα που θα μειώσουν την ψαλίδα. Διότι αυτό έχει ε, την εξής αιτία σε μεγάλο βαθμό ε, ε, η κοινωνία ανταμείβει κατά αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Όχι, αυτό θα πρέπει να διορθωθεί φέτος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, οπότε πάρα πολύ σύντομα να σας πω κάτι για τις πολλαπλές ε, διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες και ανέφερε η κυρία Σωράγια Πόστ. Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην Ευρώπη. Βλέπουμε φρικτά ε, πράγματα και καταστάσεις. Ε, συζητώ με ανθρώπους που εργάζονται στις κοινότητες Ρωμά και απευθύνομαι και στους ίδιους τους Ρωμά και τις κοινότητές τους και μας λένε ότι οι γυναίκες είναι ε, θύματα βίας ενώ φέρουν όλο ε, το βάρος της οικογένειας και επίσης πληρώνουν τους λογαριασμούς για την οικογένεια και υφίστανται και ε, κακοποίηση από εκείνους που έρχονται να ανακτήσουν τα ποσά αυτά και τους λογαριασμούς. Ε, ένα τελευταίο, περισσότερες γυναίκες σε λήψη αποφάσεων. Ξέρετε ότι προσπαθώ να προωθήσω την οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, Women on Board, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει τροποποιηθεί αυτή η οδηγία σε μεγάλο βαθμό ε, ε, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, διότι εγώ ήθελα να διατυπώσω την οδηγία αυτή ε, ουδέτερη ως προς το φύλλο, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα και ήταν αντιπαραγωγικό. Διότι το θέμα δεν είναι να αντικαταστήσουμε ε, άνδρες που έχουν πολύ ψηλά προσόντα και δεξιότητες από κάποιες γυναίκες. Όχι, θέλουμε να υπάρχει δίκαιος ε, και θεμητός ανταγωνισμός. Ε, αυτή την κατεύθυνση θα πάρει οδηγία και τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη τέτοια νομοθεσία όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία και κάποια άλλη αλλά θα χρειαστεί να μας βοηθήσουν για να φτάσουμε στα ίδια αποτελέσματα σε όλα τα κράτη. για να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στις λήψεις αποφάσεων. Αυτό δεν είναι θέμα μίας οδηγίας. Χρειάζεται νομοθεσία, χρειάζονται πολιτικές ε, σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική ζωή, γιατί έχω και κάποιες ε, επιφυλάξεις εγώ μέχρι που θα πρέπει να προχωρούμε. Αλλά αυτό αφορά γενικά το δημόσιο βίο και τις δημόσιες θέσεις, όχι μόνο στις επιχειρήσεις εταιρείες. Ξέρετε ότι είμαι και επίτροπος για τη δικαιοσύνη και στο δικαστικό. Δεν έχουμε πάρα πολλές γυναίκες σε υψηλές θέσεις ε, δικαστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσω μια, μια θετική νότα με ένα μήνυμα και προς τους άντρες. Νομίζω θα ήταν λάθος να σκέφτεστε ότι οι γυναίκες ε, θέλουν ε, να σας έχουν αντιπάλους. Όχι, συνεργάτες θέλουμε για να αλλάξουν τα πράγματα και πιο γρήγορα. Και θα χρειαστεί και η ε, συνεργασία των ανδρών, οι οποίοι κατανοούν πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη ε, μόνιμη και διαρκή προσπάθειά σας που σας υποστηρίζετε. Ε, και πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Ε,